Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Σήμερα το πρωί θα ψηφίσουμε τις πιστώσεις για τα λοιπά τμήματα τις πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις πληρωμές. Έχετε, φαντάζομαι, βάλει την κάρτα στο μηχάνημα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να κάνουμε τεστ, θα έλεγα όχι. Η πρώτη ψηφοφορία αφορά την ε, κατάσταση, την επαναφορά μάλλον, κάποιων πονδυλίων. Για να είμαστε συνεπείς, θα ξεκινήσουμε με τις πληρωμές. Για να ολοκληρώσουμε το τμήμα 3. Για τις πληρωμές λοιπόν, έχετε μία πρώτη ομάδα που τη βλέπετε αναλυτικά στο πίνακα ενός παραρτήματος. Ποιοι είστε υπέρ, ποιοι είστε αντίθετοι, ποιοι απέχουν, εγκρίνεται. Δεύτερη που για επαναφορά το πιστώσεων του σχεδίου, το βλέπετε στον πίνακα 2, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτη που Που είναι πιο ψηλά τα κονδυλιά από το σχέδιο προβλησμού. Στον πίνακα 3 βλέπετε τα σχετικά. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τέλος έχουμε την τέταρτη ομάδα πίνακας 4 στο παράρτημα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε στις χωριστές ψηφοφορίες. Συμβιβαστική τροπολογία στην υπομάδα 3, 08 080206. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία γκου 71-24 καταπίπτει. 13-03-17 τροπολογία με 90-01. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στα άλλα τμήματα. Η κεφάλαια πρώτα-πρώτα. Εδώ πρόκειται για αποκατάσταση των πιστώσεων σε σχέση με το σχέδιο του προϋπολογισμού. Προ προτάσεις ε, του Συμβουλίου και αφορά το ελληνικό συνέδριο, ε, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, την υπηρεσία προστασίας δεδομένων και άλλους οργανισμούς. σε σχέση με αυτό. Επομένω ψηφίζουμε ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνονται. Παρακάτω έχουμε τις πιστώσει του Συμβουλίου για το δεύτερο τμήμα. Έχουμε μια δέσμη τροπολογιών. Ο σκοπός είναι να περικοπούν οι πιστώσει του Συμβουλίου. Αντίθετα με τη δική μας θετική στάση ότι δηλαδή θέλαμε να ισχύσουν οι προτάσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροπολογίες μπορούν να ψηφιστούν όλες μαζί αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση. Επομένως, ποιοι είναι υπέρ αυτών των τροπολογιών. Ξεκινούν από το 1100 και φτάνουν 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 1100 έως 2237. Τέταρτο τμήμα. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κονδύλιο. 1406. Έχουμε τις τροπολογίες Γιούρι Άλντε και προϋπολογισμών. Αφορούν κάποιες επιστώσεις πέραν του σχεδίου προϋπολογισμού. 1.256.000 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κατόπιν η FDD υπάρχει αυτή η τροπολογία η οποία καταπίπτει πάμε τώρα στο 2% έχουμε τρεις τροπολογίες της Γιούρι, της Άλντε και προϋπολογισμών ούτως ώστε οι πιστώσεις να αυξηθούν πέραν της πρότασης του σχεδίου στα 659.000 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπάρχει τροπολογία των πρασίνων, η οποία όμως καταπίπτει. Γιατί εγκρίθηκε η τροπολογία αύξηση των σχετικών πιστώσεων. Τώρα έχουμε μια δέσμη τροπολογιών. Στόχος είναι η μείωση των πιστώσεων σε σχέση με το σχέδιο του προϋπολογισμού. Ξεκινούμε από το 104 και φτάνουμε στο 254 και μπορούμε, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, να τα ψηφίσουμε όλα μαζί, όλες μαζί αυτές τις τροπολογίες. Συμφωνεί και ο εισηγητής υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτονται. Παρατηρήσεις και αποθεματικά. Κονδύλι χίλια. Αμοιβέ ε, και άλλες παροχές. Μιλάει για αυτό το 3% κόντου αποθεματικό. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1400. Τροπολογία Γιούρι. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2008 Γιούρι υπέρ κατά αποχές Πέμπτο τμήμα ελεγκτικό συνέδριο Κονδυλή 1200. Υπάρχει τροπολογία εδώ της Επιτροπής Προπολογισμών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτω. Τροπολογία Σοσιαλδημοκρατών, της Άλντε και των προϋπολογισμών. επαναφέρονται οι πιστώσεις όπως προέβλεπε το σχέδιο προϋπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η τροπολογία 8.169 της FTD καταπίπτει Κονδύλι 1612 περαιτέρω κατάρτιση του προσωπικού των υπαλλήλων. Πρώτα πρώτα ε, τροπολογία της CFDD. Ο πόστοχος είναι να περικοπούν οι σχετικές πιστώσεις που είχε βασιστεί το Συμβουλίο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τέσσερις τροπολογίες σοσιαλδημοκρατών. Άλτε, Πρασίνων, και προϋπολογισμού. Ούτως ώστε να επανέλθουν οι πιστώσεις που προβλέπει το σχέδιο προπολογισμού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 162. Τροπολογία προϋπολογισμών. rétablir partiellement les crédits. Ώστε εν μέρη να επανενταχθούν στον προπολογισμό οι προβλεπτήσει πιστώσει υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Τέσσερι τώρα. Σοσιαλιστών, φιλελευθέρων, πρασίνων και προπολογισμών. το ώστε να επανέλθουν οι πιστώσεις όπως προβλέπεται το σχέδιο προπολογισμού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία της FDD καταπίπτει. 2007 Fitting out σε σχέση με τις εγκαταστάσεις. Η τροπολογία της CFDD σε σχέση με τη πιστό συμβουλίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τέσσερις τροπολογίες σοσιαλιστών φιλελευθέρων πρασίνων και προϋπολογισμών έτσι επαναφέρονται οι πιστώσεις του σχεδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 2102. Εξωτερικές υπηρεσίες για λειτουργία, εφαρμογή, συντήρηση του λειτουργικού συστημάτων και software και αυτά. Τέσσερις τροπολογίες εδώ, σοσιαλιστών, πρασίνων, φιλελευθέρων και του, της Επιτροπής του Προϋπολογισμού. Παναφορά του σχεδίου, υπέρ, κατά, α, αποχές, εγκρίνεται. 212 έπιπλα προϋπολογισμών επαναφορά εν μέρη των πιστώσεων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τέσσερις τροπολογίες σοσιαλιστών φιλελευθέρων πρασίνων και προϋπολογισμών ούτως ώστε να επαναφέρουμε τις πιστώσεις του σχέδιου προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η επόμενη τροπολογία της EFTD καταπίπτει. Κοντήλη 238 λοιπές διοικητικές δαπάνες προϋπολογισμών. 203 επαναφέρει εν μέρη τις πιστώσεις του σχεδίου προϋπολογισμού υπέρ. κατά. Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας ε, ευκρινώς. Δεν ε, καταλαβαίνω τι ψηφίζετε, άρα θα κάνουμε έλεγχο, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. πέρασα σε repoussé. Απορρίπτεται. 25-4 το σκορ. Οπότε πιο εύκολα να σηκώνετε το χέρι σας πιο ευδιάκριτα. 4. τώρα είναι η τροπολογία σοσιαλιστών, φιλελευθέρων, πρασίνων και προπολισμών, τόσο ώστε να επανέλθουν οι πιστώσεις. Υπέρ. Κατά. άποχες Εγκρίνεται. Επόμενη είναι από το EFDD, το 92 και καταπίπτει 270. Περιορισμένες διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες. Δύο τροπολογίες, ΕΛΚ και των σοσιαλιστών. Πρόκειται την αλλαγή που ήδη μας εξήγησε ο εισηγητής για το 270 αν ψηφιστεί τότε θα καταπέσουν αυτές οι όχι τότε αυτές οι τροπολογίες θα επαναφέρουν τις πιστώσεις που προβλέπονται επομένως αυτό που θα ψηφίσουμε έχει να κάνει και με τα αποθεματικά υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 2.741 τροπολογία των προϋπολογισμών για εν μέρη αποκατάσταση επαναφορά των πιστώσεων. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τέσσερις τροπολογίες σοσιαλιστών, φιλελευθέρων, πρασίνων και προϋπολογισμών. για επαναφορά των πιστώσεων του σχεδίου προπολογισμού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Και τώρα έχουμε κάποια κονδύλια. Ξεκινούν από το 2000 Από το 272. ή κάποια αύξηση σε σχέση με την πρόταση του Συμβουλίου. Αν ε, ψηφίσουμε όλες μαζί, τι λέτε. Όποιο συμφωνεί να σηκώσει το χέρι. Περ, κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Réserve, le vote a été exprimé en liaison avec... Euh, για απόφαση που έχει σχέση και με κάποιες άλλες τροπολογίες 8.028 και άλλη μία. Τώρα έχουμε το επόμενο τμήμα το οποίο αφορά την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ε, τροπολογία ENF η οποία απορρίπτεται κατόπιν της EFDD 7395 για κάποια περικοπή των όσων είχαν εγγραφεί στο σχέδιο προπολογισμού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ίντα και σοσιαλιστών. Για ε, κάποια αύξηση των πιστώσεων υπέρ κατά αποχές. Δεν μπορώ να διακρίνω ποιο σήκω στο χέρι. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τώρα ψηφίζουμε. Tout le monde a voté Il y a toujours deux parmi vous qui ne votent pas, en dépit du fait que leur carte est dans l'appareil. Eh bien, le scrutin est clos. Πέρα ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 21, 10. 1008. Η FTD. Η σχετική τροπολογία προβλέπει την περικοπή των πιστώσεων σε σχέση με το σχέδιο υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105. Κατάρτιση με τα ξενογλωσσών κλπ. Η e FDD για περικοπή των πιστώσεων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1200 αμοιβές αποζημιώσεις επιδόματα EFDD περικοπή πιστώσεων υπέρ κατά Α, αποχές απορρίπτεται. ENF 82-30. Και εδώ προτείνεται υπέρ περικοπή υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ίντα και σοσιαλιστών. Υπέρ. Κατά. Το αποτέλεσμα δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Όχι από ό,τι φαίνεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 21-9. 1220. Τροπολογία του ΙΕΝΕΦ 8231. Για απαλληφή κάποιο κοντιλίο. Απορρίπτεται. 1400. EFTD. Μείωση πιστώσεων υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1420. Πρώτον, ECR κάποια μείωση των πιστώσεων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η FTD για περικοπή των πιστώσεων υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1422 τοπολογία της EFTD περικοπή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1610 τροπολογία EFTD μείωση πιστώσεων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1612 δύο τροπολογίες του ΕΛΚ και των σοσιαλιστών για παραφορά των προβλεπωμένων πιστώσεων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 τροπολογία προϋπολογισμών για μείωση πιστώσεων υπέρ κατά σηκώστε το χέρι υπέρ είναι υπέρ της τροπολογίας 2.400 κατά αποχές απορρίπτεται 2.000 EFTD 7.406 μείωση υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2001 τι CNF 82.32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2007 προϋπολογισμών μείωση πιστώσεων. Υπέρ. Κατά. αποχές. Απορρίπτεται. 2022. EFTD. Μείωση υπέρ. Κατά. αποχές. Απορρίπτεται. Προϋπολογισμό. Μείωση πιστώσεων. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2024 τροπολογίες ECR και EFDD για μείωση υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2% EFDD μείωση πιστώσεων υπέρ κατά Α, αποχές, απορρίπτεται. Δύο τροπολογίες του ΕΛΚΑ και των σοσιαλιστών για επαναφορά των πιστώσεων. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 2.102. Η FTD, Μείωση πιστώσεων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 212 τροπολογία EFDD μείωση υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δύο τροπολογίες του ΕΛΚ και των σοσιαλιστών για επαναφορά των πιστώσεων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 214 EFDD μείωση των πιστώσεων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 216 EFDD μείωση πιστώσεων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 238 EFDD μείωση πιστώσεων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προϋπολογισμών για μείωση των πιστώσεων υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. 2540 πρώτη τροπολογία η FTD 7416 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται badge 2404 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ΕΛΚ 8032, Σοσιαλιστές 7686. Επαναφορά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 2542. Έχουμε την τροπολογία ΕΛΚ 8033, Σοσιαλιστές 7662 για επαναφορά των πιστώσεων ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε καταπίπτει του η FTD και πηγαίνουμε στην 2546 FTD 7418 για να είναι πιο μικρές πιστώσεις που αυτά προτείνουν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα έλκο 8034 και 76 776-63 για επαναφορά των πιστώσεων του σχεδίου. Περ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 2548 για το 19 FTD Περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FTT 419 Αλεξανό. Πρώτη υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. ΕΛΚ 80-35 και σοσιαλιστε 7664 Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Στο 26.00 ΕΛΚ 80-36 και σοσιαλιστε 76 76-65. Αναφορά πιστώσεων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και καταπίπτει του EFTD 7420. 2602. EFTD 7421. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2620. Ευθυντή 422 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Badge 2405. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έργο 8037 σοσιαλιστές 76-66. Με παναφορά. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26-22 γραμμή τώρα. Δύο τροπολογίε ΕΛΚ 8038, Σοσιαλιστές 7667, επαναφορά ψήφι υπέρ. Κατά, Αποχέ. εγκρίνονται. Επόμενε καταπίπτουν. Δηλαδή, ECR 8342, FTD 7423. Και στη γραμμή 2624 τώρα έχουμε την EFTD 7424 που ε, περιορίζει, μειώνει τις ε, πιστώσεις υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Πάμε στο 7ο τμήμα, Επιτροπή των Περιφερειών. Χίλια. Έχουμε τροπολογία σοσιαλιστών 77-10. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1004 ή FTD 7425 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 ΕΛΚΟ 8039 Σοσιαλιστές 7711 ψήφι υπέρ κατά δεν είναι σαφές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά και την ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Όχι από ό,τι φαίνεται. Λείπουν τρεις. Πέρασε ψηφοφορία τώρα. Εγκρίνεται. 19 υπέρ, 11 κατά και 2 αποχές. Πηγαίνουμε στο 1200. Πρώτη τροπολογία FTT 7426. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ENF 8234. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ΕΛΚ 8040. Σοσιαλιστές 7668. Παναφορά των πιστώσεων. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Καταπίπτει η μπάτζ 25.00. Στη γραμμή 12.20 έχουμε τροπολογία INF 82.35 για κατάργηση. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Στη γραμμή 1400 έχουμε την EFTD 7427 ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΕΛΚΟ 8041, Σοσιαλιστές 7669, επαναφορά. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1402. Η FTD 7428 κάτω από τις προτάσεις του Βουλιπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ΕΛΚΟ 8042, σοσιαλιστές 7670, αποκατάσταση, ε, αναφορά, πήρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1420, FTD 7429, κάτω από το σχέδιο του προπλήρου, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται ελκε 8043, 80-43, σοσιαλιστές 12 Πάνω από το σχέδιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 1422. Η FTD 7430. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16-10. EFTD 74-31. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16-12. EFTD 74-32. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπάτζ 25-01. Διαπιστώσει κάτω από το σχέδιο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 162 ECR 83-32. Κάτω του σχεδίου Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλκο 80-44, σοσιαλιστές 76-87. Πάνω από το σχέδιο Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2000. EFTD 7434 Κάτω από το σχέδιο προπολογισμού. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 2007 έχουμε 8045 και σοσιαλιστες 7688 για αύξηση σχέση με το σχέδιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Και επόμενη, μπάτζ 2502, καταπίπτει. Στο 2022 έχουμε το FTD 7435, μείωση σε σχέση με τις προβλέψεις του Συμβουλίου. κατά, αποχές, απορρίπτεται, έλικο 8047 και σοσιαλιστές 13 για επαναφορά. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Καταπίπτει η μπάτση 2503. Πάμε στο 2024. Έχουμε την EFTD 7436. Μείωση σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στο 2100 έχουμε την ΕΛΚΟ 8048 και την Σοσιαλιστό 7689 αύξηση. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει επόμενη. 2102. Έχουμε την EFTD 7437. Μείωση σε σχέση με το σχέδιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 212. EFTD 7438. Μείωση. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στο 2.14 την e FTD 74.39 για μείωση. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε την ΕΛΚΟ 8046 και στους 7690 για αύξηση. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και επομένως καταπίπτει επόμενη. Μπάτζ 2505. 216. Η FTD 7440 για μείωση. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 2.30. FTD 7441. Μείωση. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.38. FTD 7442. Μείωση. Ψήφι υπέρ. Κατά. Α... Ορίστε. Εκτός μικροφώνου όχι δεν γίνεται. Συγγνώμη. Άρα απορρίπτεται. Έχουμε την AFTD 7443 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Στο 2541 FTD 7444 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2542 FTD 7445 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Badge 2506 υπέρ για μείωση υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 2546 FTD 7446 μείωση υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 2600 FTD 7447 μείωση υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Badge 2507 μείωση υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 2602. Μπάτζ. 2508. Μείωση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2620. 8049. Ε, σοσιαλιστές. 7708. Επαναφορά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι δύο επόμενες. 2622. Σοσιαλιστές 7714. Αύξηση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και η FTD 7449 καταπίπτει. 264 ΕΛΚ 8050 και Σοσιαλιστές 7709. Αύξηση. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και το ECR 8333 καταπιπτει πίπτη. τμήμα τώρα για το διαμεσολαβητή. Εδώ νομίζω μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες από την 104 στην 303. Τι λέει ο συγητής μας, συμφωνεί. Άρα Ποιοι είναι παρακαλώ υπέρ των έξι αυτών τροπολογιών. Σηκώστε τα χέρια σας. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν παρακαλώ. Απορρίπτονται οι τροπολογίες αυτές. Πηγαίνουμε στο ένα το τμήμα που είναι επόπτης προστασίας δεδομένων. Νομίζω και εδώ μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού τις τροπολογίες από το 10-10 έως το 3044. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, σκώστε τα χέρια, κατά, αποχές, απορρίπτονται οι τροπολογίες αυτές. 10, τμήμα 10. Η ΑΕΔ, περί εξωτερική δράση. Στο 1200 Έχουμε την τροπολογία ΑΦΕΤ 5306 για αύξηση. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και οι επόμενες 3, η ΕΝΕΦ 8242, FTD 8554, ECR 8330 καταπίπτουν. 2214. Νέα. Νέο κονδύλιο. ΑΦΕΤ 5221, BADGE 4408. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 30.02 η πρώτη τροπολογία 52.60. Αύξηση. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το INF 8292 και το FTT 8558 καταπίπτουν. Στο 3006 έχουμε την ΑΦΕΤ 5308. Α, δεν πρέπει να ψηφιστούν αυτές. Άλλα τώρα κονδύλια στο 1101. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα ψηφίσουμε από κοινού και να πάμε μέχρι πού. 3005. Συμφωνεί ο συγγητής. Συμφωνεί. Lequel celui-là Le budget 40. Bon, alors, on va voter, on va voter. Donc on va, monsieur... Λοιπόν, ο κύριος Ρούμπικ θέλει να ψηφίσουν τροπολογία του badge 4625. Άρα θα έχουμε ένα πρώτο μπλοκ από το 1101 έως το 1202. Σε το συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, μέχρι το 12.01, τρεις τροπολογίες δηλαδή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι τρεις πρώτες τροπολογίες απορρίπτονται στο 12.02. Έχουμε την τροπολογία ΙΕΝΕΦ καταρχάς, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και έχουμε τη δεύτερη τροπολογία Μπατζ, 4625 του κ. Ρούμπιχ τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. 22 κατά, 12 υπέρ, άρα απορρίπτεται. Και αν συμφωνεί τώρα ο μπορούν το 1203 μέχρι το 3005 να ψηφίσουμε από κοινού αν συμφωνείτε. συμφωνείτε. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν αυτή της τροπολογιών. Ποιοι είναι κατά. Και απέχουν. Απορρίπτονται αυτές τις τροπολογίες. Και φτάνουμε στις παρατηρήσεις. Στο 1200. Άφετ 5306. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στο 30.02 άφετ. 52.60 ε, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30.06 άφετ 53.08 ΕΛΚ 80.27 μπατ 46.08 Δεν χρειάζεται να τις ψηφίσουμε που σημαίνει ότι πηγαίνουμε στο τμήμα 1. Δηλαδή, στον προεπλισμό του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, έχουμε μια πρώτη ψηφοφορία για τη διατήρηση των πιστώσεων. Με το ντοκιμαντέρ της του τα βλέπω στο παράρτημα πίνακα 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές γκρίνεται. δεύτερη ομάδα της λεπτομέρειας των πίνακα 2, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και έχουμε κάποια νέα αιτήματα. Στο 1200 κοντήλι, τροπολογία Γκουε, 7313. για αύξηση. Όχι, για μείωση. Τέλο πάντων, μπορούμε να τα ψηφίσουμε μαζί και τα δύο γιατί σχετίζονται το ένα με το άλλο. Μεταφορά πιστώσεων είναι. Για διοικητικού μισθού προ ομάδε. Ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές οι διατροπολογίες. τροπολογίες. 73-13-73-14 της ΓΚΟΕ. Έχουμε τώρα στο 1006 να ψηφίσουμε την badge 46 για το απόθεμα. 10% περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και πηγαίνουμε στις παρατηρήσεις. Στο κοντιλί 242 έχουμε την τροπολογία της ΑΦΚΟ 6736. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Θα έλεγα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 ήταν αντίθετη, 16 πέρ. Πάμε τώρα στο 3245 45 6742. πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στο 326 έχουμε την μπάζ 4627. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και το Establishment Plan στο τέλος που έχουμε το S1-12 ή FTD-86-60. Μια δραστική ε, τοποθέτηση, προσέγγιση σε σχέση με το προσωπικό των ομάδων. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Απορρίπτεται τροπολογία. Eh bien, mes chers collègues, nous en avons terminé. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε την εξέταση και την ψήφιση των τροπολογιών για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2018. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ νέου και να συγχαρώ τους εισηγητές μας, Ζίγκριτ Μούρεσαν και Ρίτσαρντ Άσχορτ. Καταπληκτική δουλειά τους διαφώτισαν την Επιτροπή Προπολογισμών. Βέβαια, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τους συνεργάτες μας. Η διάρκεια της ψηφοφορία ήταν μικρότερη από ό,τι συνήθως. Ελπίζω να μην σας δημιούργησε αυτό κάποιο πρόβλημα. Και η σύντομη διάρκεια οφείλεται στο έργο των εισηγητών, των σκιωδών εισηγητών, των πολιτικών συμβούλων, της γραμματείας που τα πήγε περίφημα και θέλω να τους χειροκροτήσουμε. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Πρόεδρο έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και χαιρόμαστε για το πώς ε, την έκανε και εύχομαι την επόμενη φορά ε, όταν ψηφίζουμε να ξέρουμε πότε ψηφίζουμε και να είναι ξεκάθαρο να ψηφίζουμε με τη μία γιατί χάσαμε σήμερα τη συνεδρία των ομάδων που πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Λάβετε λοιπόν υπόψη ε, τις απαιτήσει Θέλω πάντως να σας ευχαριστήσω. Πολύ καλή ψηφοφορία και ελπίζω η συνδιαλλαγή να έχει καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Déjà, d'ores et déjà, euh, je voudrais vous dire qu'il serait bon et sage de réserver. Το πιο σωστό θα ήταν την τελευταία τρίτη και τελευταία τετάρτη του Σεπτεμβρίου του 2018 να τις κρατήσετε για να ε, ψηφίσουμε τους, τους, για τον προϋπολογισμό του 19 και τις πολιτικές ομάδες να τις επηρεάσετε, να τους πείσετε ότι οι ψηφοφορίες για τις τροπολογίες του υπολογισμού είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Να μας πάρουν στα σοβαρά και να μας φέρονται σωστά οι πολιτικές ομάδες. Τάραντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρά το ότι χάσαμε τις ψηφοφορίες όλες, συμφωνώ με τον ε, κύριο Ρουμπιχέ. Je voudrais vous indiquer que la Commission des budgets... Ε, επίσης, η Επιτροπή Προεπολογισμών ενέκρινε τις τροπολογίες για τη χρήση του 18 και θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κύριο Ζωάν Ρέλ, διευθυντής. Μήπως έχετε κάποιες παρατηρήσεις, κύριε. Uh, for... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που μας δώσετε τον λόγο. Είμαι σύντομος. Ε, δεν ε, θα γρηγορήσω να συγχαρώ και εγώ τους εισηγητές ε, για το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα και την ψηφοφορία. Και ευχαριστώ για τη δουλειά που έκαναν ε, με την αντιμετώπιση όλων αυτών των τροπολογιών και για το ότι καταλήξαμε σε ένα επιτυχή συμβασμό. Δεν θα κάνω συγκεκριμένα σχόλια σήμερα. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν θα σα στείλει όπως κάθε χρόνο την επιστολή εκτελεστικότητας για τις λεπτομέρειες της θέσης Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Λίγα σχόλια λοιπόν σήμερα. Σε γενικές γραμμές ευχαριστούμε την Επιτροπή που ψήφισε τις ε, διάφορες ε, τροπολογίες που αποκατέστησαν το σχέδιο προϋπολογισμού. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Όσον αφορά τον τίτλο 1α θα ήθελα να εκφράσω μία ανησυχία που σχετίζεται με το ότι αφαιρέθηκαν τα κονδύλια για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και αντιλαμβάνομαι βεβαίως το σκεπτικό δηλαδή να μην προδικάσουμε την ε, νομοθετική διαδικασία, απλά έχουμε την ανησυχία ότι μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής ε, διαδικασίας με το να έχουμε βγάλει τα κονδύλια από τον προϋπολογισμό θα είμαστε αναγκασμένοι να φέρουμε διορθωτικό προϋπολογισμό που θα προκαλέσει καθυστερήσεις και θα μειώσει τις ε, δυνατότητες κινητικότητας ε, για τους νέους. Όσον αφορά τον τίτλο 1β, ένα σχόλιο μόνο για την απασχόληση των νέων. Στο σχέδιο προπολογισμού η Κομισιόν είχε προτείνει να μοιραστούν εξίσου τα ποσά που είχε συμφωνήσει Συμβουλή και Κοινοβούλιο στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση στα έτη 18-19-20. Γνωρίζω τώρα ότι υπάρχει η επιθυμία του Κοινοβουλίου τα ποσά αυτά να πάνε όλα στο 2018 να ε, μπροστοβαρείς ε, η εκταμίευση, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότερα λεφτά για το 19 και το 20. Για τον τίτλο 2, να υπενθυμίσω στους βουλευτές ότι όπως ε, κάθε χρόνο η Κομισιόν θα υποβάλει μια διορθωτική επιστολή μέσα Οκτωβρίου. Κάτι το οποίο θα σας ε, δώσει τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις. Για τίτλους 3, 4 και 5 δεν θα κάνω σχόλια σήμερα, εκτός από μία παρατήρηση. Να σημειώσουμε ένα σημείο συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, δηλαδή την επιθυμία να μειωθούν οι προενταξιακές, η προενταξιακή χρηματοδότηση για την Τουρκία. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Ευχαριστώ λοιπόν που μου δώσατε τον λόγο τη χαρτίρια στους και αναμένουμε μια εξίσου επιτυχημένη ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου και νομίζω τώρα έχουμε μια πολύ καλή βάση για να πάμε στην συνδιαλλαγή. Για να ολοκληρωθεί ε, επιτυχώ ο προπολογισμό του 2018. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Διευθύντα για τα σχόλιά σα τα οποία σημειώσαμε. Σας ευχαριστώ και για τις ε, επικοδομητικές σχέσεις που έχουμε με την Κομισιόν και ειδικά τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού. Κύριε Ισηγητά, θα θέλατε να μας πείτε κι εσείς πώς νιώθετε μετά από όλη αυτή τη διαδικασία. Κύριε Μουρεσάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν παρόντες ε, και χτες και σήμερα. Νομίζω είναι σαφές ε, το μήνυμα προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο ότι προετοιμάζουμε εξαντλητικά την θέση του Κοινοβουλίου όλα τα σημαντικά στοιχεία ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν και ψηφίστηκαν και ελπίζω ότι το ίδιο θα κάνει και η Ολομέλεια στο τέλος του Οκτωβρίου και ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την θέση του Κοινοβουλίου. Για την Κομισιόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια που κάνατε. Αναφέρατε και πριν το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού στο πλαίσιο του τίτλου 2. Βεβαίω είναι συνήθι διαδικασία, αλλά βεβαίω γνωρίζουμε ότι η τροποποιητική επιστολή πιθανότατα θα πάει πέρα από τον τίτλο 2, γιατί είναι βεβαίω και λύπηρο το ότι δεν ενημερώθηκε πιο λεπτομερό το Κοινοβούλιο για την τροποποιητική επιστολή, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ε, θα είχαμε διαφορετική κατάσταση. Αν υπήρχε βεβαίως μεγαλύτερη διαφάνεια και γνωρίζαμε τα πράγματα, ε, θα τα είχαμε λάβει υπόψη στην ψηφοφορία. Τώρα είμαστε σε μια θέση όπου έχει μια ξεκάθαρη θέση το Κοινοβούλιο και βεβαίως ε, το θέμα αυτό το οποίο πρέπει να μεταφέρετε στον Επίτροπο τον κύριο Έτιγκερ είναι ότι θα είναι δύσκολη η συνδιαλλαγή εάν η Κομισιόν επιλέξει να μην λάβει υπόψη την θέση του Κοινοβουλίου όταν θα παρουσιάσει την τροποποιητική επιστολή. Οπότε, όσα περισσότερα βάζουμε, όσα περισσότερα δεχτείτε και βάλετε στην επιστολή σας από αυτά τα οποία ψήσαμε χθες και σήμερα, τόσο ευκολότερα θα είναι τα πράγματα και βεβαίως ε, η συνδελεγή γίνεται έτσι κάπως πιο εύκολα και για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ε, η αύξηση προτείνουμε δεν είναι κάποιου είδους εμπροστοβαρής εκταμίευση είναι απλά να προτείνουμε μια αύξηση για να αντιμετωπίσουμε την πολύ υψηλή ανεργία των νέων στα κράτη-μέλη και θεωρούμε ότι το ποσό το οποίο προτείνει η Κομισιόν 233 εκατομμύρια ευρώ δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσουμε το μέγεθος της πρόκλησης. Θεωρούμε απλά ότι απαιτούνται περισσότερα κονδυλία. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε εδώ πέρα και ψηφίζετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γενικό Συγητή και τώρα ο κύριος Άσουερθ θα πάρει το λόγο που έκανε και αυτός καταπληκτική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την βοήθεια, την υποστήριξη, να βοηθήσω και τους σκιώδους για τη δική τους δουλειά για τον προπολογισμό αυτό. Όπως είπα και ευθύ εξ αρχής το Κοινοβούλιο είχε βάλει αύξηση 2,3% πέρυσι για τον προπολογισμό. Θεωρούσα ανέκαθεν εγώ ότι αυτό ήταν ε, ένα όριο αναφοράς λογικό και θα ήταν και η βάση σύγκριση με τα άλλα θεσμικά όργανα. Έλεγα βέβαια ότι αυτό σημαίνει ε, πειθαρχία και δύσκολες αποφάσεις και είναι σαφές απορισμένο. Στις ψηφοφορίες ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν συμφωνούν μαζί μου και θα τη σεβαστώ την απόφασή τους ο προπολογισμό, δεν ξέρω ακριβώ ποιο θα είναι το ποσοστό, θα είναι πάντω αυξημένο γύρω στο 3%. Σέβομαι τις απόψεις παρότι δεν είμαι απόλυτα προσωπικά. Το έγγραφο που έχουμε πάντως νομίζω ότι μπορούμε να το υποστηρίξουμε στις ε, διαδικασία συνδιαλλαγής με Συμβούλιο και Κομισιόν και ελπίζω να στεφθεί με επιτυχία η διαδικασία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρία Σουέρθ. Και εκτιμώ το ότι θέλατε να είστε οικονόμος με τα δημόσια κονδύλια. Και πράγματι. Πήραμε κάποιες δεσμεύσεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τη συνδιαλλαγή μπορεί να μας τις περικόψουν τις φιλοδοξίες μας στη συνδιαλλαγή. Ο Ζήκερ Ρεκμούρεσαν μίλησε για τους νέους, για την απασχόληση των νέων. Αν με επιτρέπετε μια προσωπική παρατήρηση, αρκετοί από εμά έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο πιλωτικό, ώστε οι μαθητευόμενοι να παίρνουν, ε, να, να από το Εράσμους για την κινητικότητα. Ο πολιτισμός ε, για χώρες όπως Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία που έχουν κάποια τέτοια προγράμματα είναι κάτι θετικό και με τον τρόπο αυτό υπάρχει πιο μεγάλη ένταξη. Η Κομισιόν το συμπεριέλαβε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα στο πρόγραμμά της. 400 εκατομμύρια θα είναι ο προπολογισμό για τις υποτροφίες Εράσμους, για τους μαθητευόμενους, για τους ασκούμενους. Και πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ θετικό για να κάνουμε τους νέους να νιώσουν Ευρωπαίοι πιο πολύ, να βρουν επίσης μια θέση εργασίας. Και επειδή 28 χώρες είναι 28 διαφορετικές νομοθεσίες, πρέπει να έχουν υπόψη ότι θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις στις κυβερνήσεις για να αλλάξουν την νομοθεσία τους και να προχωρήσουμε ίσως προς ένα νέο πλαίσιο σε ό,τι αφορά το καθεστώς του ασκούμενου στην Ευρώπη. Πολύ προσωπική παρατήρηση και πριν κήρυξω τη λήξη της συνεδρίασης να σας πενθυμίσω ποια είναι τα επόμενα στάδια. Θα ψηφίσουμε το ψήφισμα της δημοσιονομικές τροποποίησης στις 10 Οκτωβρίου Επιτροπή Προϋπολογισμών, τριμερής διάλογος, πρώτος 18 Οκτωβρίου, συζήτηση και έγκριση στην Ολομέλεια της θέσης του Κοινοβουλίου 24-25 Οκτωβρίου, και η περίοδος συνδιαλλαγής. Θα ξεκινήσουμε πρώτη συνεδρίαση στις 6 Νοεμβρίου, δεύτερη, ελπίζουμε και τελευταία, στις 17 Νοεμβρίου. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τη συνδιαλλαγή, αν θέλουμε ένα θετικό το αποτέλεσμα, πριν τις 20 Νοεμβρίου. Με αυτά και με αυτά έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις στα διάφορα κάτι, αν όχι κηρύσω τη λήξη της συνεδρίασης.